Πολύ ε, να συμφωνήσουμε με αυτά τα οποία έγιναν ε, χθε και αυτά που είπε ο πρόεδρος Σούτς επομένω σε σχέση με τον συνάδελφο Μπονάνο ο οποίος ε, πέθανε κατόπιν ενός αυτοκινητικού ατυχήματος και επομένω στα συλληπιτριά μας στην οικογένειά του, στους φίλους του αλλά βέβαια και στην πολιτική ομάδα στην οποία ανήκε. Έχουμε και κάποια άλλη ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές της Σουηδίας επικοινώνησαν με τον ε, πρόεδρο και ανακοίνωσαν την εκλογή του κυρίου Γιάκοπ Νταλόντε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον κύριο Πίτερ Έριξον, κάτι το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από τις 7 έκτου του 16. Καλώς όρισε ο νέος συνάδελφος και σας υπενθυμίζω ότι θα είναι πλήρως ε, μέλος του Κοινοβουλίου και θα συμμετάσχει σε τον κανονισμό σε όλα τα όργανα του Κοινοβουλίου μας. Και τώρα οι ψηφοφορίες που προβλέπουν